Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι τρεις και δύο λεπτά και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε λάβει όλη την εμείς διάταξη, νομίζω μπορούμε λοιπόν να την εγκρίνουμε. Το σημείο 2 τώρα, οι ανακοινώσει του Πρόεδρου, να σας ενημερώσω ότι ο συνάδελφος μέλος της ΙΝΤΑ και ε, συντονιστής ο Εντουάρ Φερό μας άφησε την 1η Φεβρουαρίου του 2018. Ήταν μέλος από το 2015 του Κοινοβουλίου και βεβαίως στα θερμά μου συλληπιτήρια στους συναδέλφους, στην οικογένεια. Ένα λόγο από τους θα σας ζητήσω. Η πρώτη ανακοίνωση είναι ότι αυτή η συνάντηση βεβαίως ως συνήθως μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Υπάρχει διερμηνία. Μιλήστε λοιπόν δυνατά και καθαρά για να βοηθήσετε το έργο των διερμηνέων. Για τους ε, προσκεκλημένους μας ε, επίσης να κάνετε μια προσπάθεια να σας πω επίσης ότι έχουμε ένα νέο συνάδελφο τη Μόνικα Μίγκο που δουλεύει εδώ και καιρό βεβαίως στην γραμματεία ατύπως αλλά πλέον αναλαμβάνει και επισήμως. Point uh, Σημείο 3 τώρα. Αποκινούμε την ε, Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, θα εξετάσουμε το σημείο αυτό. Ε, ορίζω την εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής ΔΕΒΕ, την πρώτη Επιτροπής ΔΕΒΕ. Θα θυμάστε ότι προέκυψε μια πολύ καλή ε, νομοθεσία για τα ορυκτά στις περιοχές σειράξεων ξέρουμε ότι αυτή η νομοθεσία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά από τέσσερα χρόνια από την 1η του 2021. Υπάρχει δηλαδή μια μεταβατική περίοδο μέχρι τότε, μεγάλη μεταβατική περίοδο, αλλά από την άλλη ε, μπορέσαμε να περάσουμε πολλά σημαντικά ζητήματα μέσω αυτή τη νομοθεσία. Βεβαίω ε, η νομοθεσία είναι, μέρο, είναι, το ένα μέρο ε, του όλου ζητήματο. Υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος όμως. Το θέμα είναι πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση επιτόπου πώς θα προετοιμάσουμε αυτή την ενίσχυση με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγυηθεί ότι μαζί με την εφαρμογή της νομοθεσίας, η διαδικασία εφαρμογής θα πρέπει να οργανωθεί σωστά και να παρακολουθείτε. Αυτό είναι το θέμα που θα μας προσχολήσει σήμερα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ Μπέρντ και ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να έχουμε μια κοινή συζήτηση των δύο επιτροπών. Όπως είπατε, μιλάμε για τα ρηκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και το θέμα είναι ε, να μην έχουμε μόνο τις νομοθετικές διατάξεις αλλά και συνοδευτικά μέτρα για την εφαρμογή αυτών των νομοθετικών διατάξεων. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της μιλούσε για αυτά τα συνοδευτικά μέτρα του κανονισμού αλλά αυτό ήταν πολύ, έγινε παλιά, πριν από τρία χρόνια. Ε, ήμουν ακόμη τότε πρόεδρος της Επιτροπής και ενώ έχουν περάσει τρία χρόνια, το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε κάποιες προτάσεις ε, για 4,5 εκατομμύρια για το, ε, για το κοινό αυτό πρόγραμμα για τα δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις με συνδιαχείριση μιας ε, Ολλανδικής εταιρεία, του Ολλανδικού Οργανισμού Επιχειρήσεων. δεν ξέρω αν θεωρεί ότι εξαντλούνται εκεί οι ε, νομοθετικές υποχρεώσεις ή θα πρέπει να προτείνει και άλλα συνοδευτικά μέτρα για να ευοδοθεί η εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια σχετική συνάντηση και θέλουμε το θέμα των ορεικτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ευχαριστώ ε, τον Μπέντ και την Επιτροπή ΝΙΤΑ που είναι η κυρία Σαρμόδια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές, από την Ίντα στον κύριο Βίνκλερ και από την Τέβε στον κύριο Βέντα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε και θυμόμαστε, έχει γίνει μεγάλη προεργασία από τους συνεισηγητές, τους και ε, και της ε, γραμματείας των δύο επιτροπών. Θα θυμάστε ότι τον Ιούλιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2017 υπεγράφει ο κανονισμός και τέθηκε σε ισχύ και Έχουμε τώρα κάποια χρόνια μέχρι την ε, οριστική θέση εφαρμογή μετά τη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει τώρα να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό με μεγάλη περιέργεια περιμένουμε τα κέρια αυτά σημεία, τα βασικά σημεία. Καταρχήν σημειώθηκε κάποια πρόοδος ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους διάφορους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικούς τελεστές επιχειρήσεις και τα λοιπά εισαγωγής είναι ένα σημαντικό θέμα. Και δεύτερο θέμα είναι ε, το καθεστώς για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Καταρχήν υπάρχουν ήδη έτοιμες τέτοιες αρμόδιες αρχές. Τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Και υπάρχει δυνατότητα ή έχει τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει να συνδράμει αυτές τις συνασταθήσεις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη. Και επίσης στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, στην ΙΝΤΑ δηλαδή την Επιτροπή μας, ε, ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μικρότεροι φορείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συνεπικουρηθούν στις προσπάθειές τους να τηρήσουν αυτή την υποχρέωση δέωσης επιμέλειας που προβλέπει ο κανονισμός. Ως προς αυτό λοιπόν το θέμα υπάρχουν νέα στοιχεία. Πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επίσης, ε, ζητήσαμε να γίνουν κάποιες προσπάθειες για τη μετάφραση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΣΑ ώστε να έχουν επίσης όρις πρόσβαση σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί όπως γνωρίζουμε η, πολυγλωσ... η πολυγλωσία είναι μίζωνα πρόκληση για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, για τους υπόλοιπους εταίρους μας παγκοσμίως, Ε, ποιες είναι οι αντιδράσεις τους ε, δείχνουν κάποια δείγματα γραφής για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον κανονισμό για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, γιατί αυτός ο κανονισμός διαφέρει παρασάγκας από τις αντίστοιχες δράσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα αυτό, που προηγούνται κιόλα. Επίσης, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για την ε, πρόορη επικαιροποίηση για τους διάφορους ε, τελεστές, γιατί το 2016 και 2017 είχαν αναλυφθεί κάποιες ε, αγαστές πρωτοβουλίες για ΣΔΙΤ και άλλες συνεργασίες. Υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό. Γιατί πιστεύω ότι από κοινού με τους οικονομικούς τελεστές ε, και σε συνεργασία μόνο μπορούμε να στέψουμε με επιτυχία τις κοινέ μας προσπάθειες. Ευχαριστώ κύριος Βέντα. Ευχαριστώ. Φυσικά ο κανονισμός αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μέσο άσκηση εμπορικής πολιτικής, θα πρέπει να θεωρηθεί υπό ένα ευρύτερο ε, πρίσμα και υπό το πρίσμα της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας. Και για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του κανονισμού αυτού, ε, θεωρώ και είναι σημασίες για μένα που είμαι συγκεκριτή, της Επιτροπής ΔΕΒΕ, τα συνοδευτικά μέτρα να εφαρμοστούν εκ παραλίλου με τον κυρίως κανονισμό. Η ανακοίνωση του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε κάποια συνοδευτικά μέτρα για να ενθαρρύνει την υπεύθυνη αγορά τέτοιων ε, ορυκτών που αναφέρονται στους πέντε τίτλους. Και το 2017 πρότεινε ε, το πρώτο τέτοιο μέσο ε, αναπτυξιακής συνεργασίας με τα συνοδευτικά μέτρα, εξασφαλίζοντας υπευθυνότητα στον τρόπο αγορά τέτοιων ορεικτών. Βέβαια αυτά τα συνοδευτικά μέτρα καλύπτουν μέχρι στιγμής μόνο ένα τμήμα από τις, τους 14 τομείς εργασιών που απαριθμούνται στην αρχική ανακοίνωση του 2014. Οπότε ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτίθεται να προτείνει και συμπληρωματικά συνοδευτικά μέτρα που θα καλύπτουν και τους υπόλοιπους τομείς ε, της ανακοίνωσης θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα και προπολογισμό για όλες αυτές τις συνοδευτικές δράσεις, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές για μας. Και θεωρώ ότι είναι ε, σημαντικό να γνωρίζουμε τις προθέσεις και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ε, ε, θα χρηματοδοτηθούν και άλλα συνοδευτικά μέτρα από το σχετικό μέσο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και στην έγκριση και εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων. Γι' αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται όντω να εμπλέξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων. Αυτά και ευχαριστώ και τον Προτέρα για τι απαντήσει. Τρει συνάδελφοι τρεις μάλλον ε, εκπρόσωποι ζήτησαν το λόγο από την ε, DigiTrade, την DigiDefco και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θα ξεκινήσουμε από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. κύριος, η κυρία Ράτσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε σε αυτή τη συζήτηση. Και επίσης να σας ευχαριστήσω που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία να τεθούν προφορικές ερωτήσεις επ' αυτού του τόσο σημαντικού θέματος. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν επιδιώκει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να διασφαλίσει την υπεύθυνη εκμετάλλευση αυτών των ε, ορυκτών. Ο κανονισμός που και πέρυσι, είναι ε, ορόσημο και επειδή ε, αναφέρθηκε ήδη, θέλω και εγώ να πω ότι θα έχουμε μη ρυθμιστικά συνοδευτικά μέτρα για να στηρίξουν αυτή την προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται ολοταχώς ε, στο να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα μέσω συνεργασίας ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα τώρα εγώ, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι από άλλες διευθύνσεις που θα εκφράσουν και εκείνη την άποψη ε, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο κανονισμός ε, που τέθηκε σε εφαρμογή τέθηκε πριν από έξι μήνες. Ως εκ τούτου οι απαιτήσει ε, για τις εταιρείε θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Ως εκ τούτου εξορισμού πολλά από αυτά τα μέτρα βρίσκονται ακόμα σε προκαταρκτική φάση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ε, που να αφορούν ε, σε κάθε ένα από τα συνοδευτικά μέτρα γιατί κάτι τέτοιο κατ' ουσίαν αφορά την Ολομέλεια του Μαρτίου όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να τοποθετηθεί επίσημα στις προφορικές σας ερωτήσεις αλλά θα σας δώσω έτσι μια γενική επισκόπηση επί των θεμάτων που ανέφερε και ο Πρόεδρος αλλά και οι συγητές. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχει μια σειρά προκατρακτικών δράσεων που καθορίζονται με απόλυτη σαφήνεια στον κανονισμό και υπενθυμίζω περιλαμβάνεται, ε, περιλαμβάνονται κατευθυντήρες γραμμές ε, για το τι πρέπει να κάνουν με περιοχές υψηλού κινδύνου, ε, κατευθυντήρες γραμμές για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σχετικά με τους ελέγχους στους εισαγωγείς, λεπτομερείς διατάξεις για τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για να εντοπίζονται θέματα που έχουν σχέση με τη δέους επιμέλεια. Σε όλα αυτά έχουμε προχωρήσει. Υπάρχουν και άλλα συνοδευτικά μέτρα που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από την τελική μορφή που θα λάβουν τα προαναφερθέντα. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν αργότερα. Ε, εξάλλου, προχωράμε και γενικότερα στα συνοδευτικά μέτρα. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που έχουν σχέση με την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μέτρα που έχουν σχέση με τη δέος επιμέλεια στο κύριο κομμάτι για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Βίνκλα όσον αφορά τη μετάφραση ε, του οδηγού που έχει εκδώσει ο ΩΣΑ. Η μετάφραση είναι έτοιμη περίπου στις αρχές Απριλίου για να ε, βοηθηθούν με τον τρόπο αυτό και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί επίση ε, να υπογραμμίσει τη σημαντική δουλειά που κάνουμε με το να ενθαρρύνουμε τρίτες χώρες να παράγουν και να καταναλώνουν, να εφαρμόζουν ε, πολιτικές που έχουν σχέση με την υπεύθυνη εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών και με βάση τις κατευθυντικές γραμμές του ΟΣΑ. Ένας συνάδελφός μου από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα μιλήσει ε, και για τη ε, διαδικασία που ακολουθείται στον Όσα, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη επευθυνθεί σε μία σειρά χωρών οι οποίες και παράγουν Αναφέρομαι στι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, στον Καναδά, στην Ινδία, Νότια Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στη Μαλισία και στην Ταϊλάνδη. Και ελπίζω να μην ξέχασα καμία. Ορισμένες εξ αυτών ε, έχουν βεβαιωθεί τη δική τους τη στάση έναντι τις ε, θέσεις του ΟΣΑ, παραδείγματος χάρη η Κίνα. Αλλά ε, έχοντας κατά νου βεβαίως την προφορική ερώτηση, αργότερα θα σας δώσουμε περισσότερες ε, λεπτομέρειες από αυτού. Και θα ήθελα τώρα να μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο σε ένα συνάδελφό μου από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ο οποίος ασχολείται με ε, προγράμματα τα οποία πραγματικά ε, θα σημάνουν και μια ουσιαστική διαφορά στην πράξη. Καλησπέρα σας. Ε, να συμπληρώσω λιγάκι στα συνοδευτικά μέτρα που ανέφερε και η κυρία Μακάβεν. Πριν από κάποιους μήνες, το Δεκέμβρη, εγκρίναμε το θεματικό πρόγραμμα που αφορά ε, στις, ε, στα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 5,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, αυτές αναφέρονται στην ανακοίνωση του 2014, η ανακοίνωση εκείνη που αφορά στην ε, υπεύθυνη εκμετάλλευση ορυκτών σε περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι και οι πληθυσμοί που ζουν σε αυτές τις ε, περιοχές. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι μικρές δράσεις. Θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί η οδηγία του ΩΣΑ σχετικά με τη δέωση επιμέλεια και κυρίως τον να υπάρχουν οικονομικές ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις. Να μπορούν ε, με τα προγράμματα της δέουσας επιμέλειας να στηριχτούν η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία των πολιτών και οι μικροί επιχειρηματίες. Το να βελτιωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες αυτών των κοινοτήτων, αυτό θα περιορίσει την ε, κατάχρηση και παραβίαση των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα δώσει και τη δυνατότητα και αυτοί να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δάνεια αυτά όλα εντάσσονται στο πρόγραμμά μας των εξωτερικών επενδύσεων και κυρίως τον τρίτο πυλώνα ε, Αντιμετωπίζεις λοιπόν τις ε, άτυπες, τα άτυπα στοιχεία και την διαχείριση θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προσφέρουμε περισσότερα οικονομικά ωφέλη στις οικονομίες των λόγω κρατών. Ασχολούμεται επίσης με την υπεύθυνη εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών, τη σωστή τους εξόριξη. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και να βοηθήσουμε και τους ε, ε, φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνονται σε θέματα ε, δέουσας επιμέλειας γιατί θα υπάρχει πιστοποίηση και αυτό με βάση τις κατευθυντής γραμμές του ΟΣΑ. Όσον αφορά τώρα ε, το πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε πέρσι. Αυτή τη στιγμή συντάσσονται οι συμβάσεις και το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την υπεύθυνη χρήση ορυκτών. Πρόσφατα προέκυψε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία των πολιτών, με τους δωρητές, ε, για να στηρίξουν όλη αυτή την εφαρμογή του κανονισμού για ορυκτά σε περιοχές συγκρούσεων. Με τον τρόπο αυτό νομίζω θα βοηθήσουμε την συνεργασία ανάμεσα τους φορείς, ε, κυρίως ε, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε να εξορίσετε ε, χρυσός από περιοχές όπου δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Στην Κολομβία ε, θα μπορούμε και εκεί να εφαρμόσουμε σε όλη την αλυσίδα τις οδηγίες ε, του ΩΣΑ. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές αρχές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν αιτήσει στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Επειδή όμως το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα στην τελική του φάση, ελπίζουμε η χρηματοδότηση της πρώτης σειράς εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, διαφόρων μορφών εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτά έχουν σχέση με τον κανονισμό και νομίζω ότι ε, και εμείς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τον ΩΣΑ έτσι ώστε η δέουσα επιμέλεια να γίνεται σεβαστή, να υπάρχει γεωγραφική χρηματοδότηση μέχρι και 10 εκατομμύρια ευρώ, ευρώ. Μιλάμε για ένα σύνολο της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότηση. Αυτά είναι και η απάντηση στην επιστολή που στάλει πριν από τρία χρόνια ε, σε διάφορες επιτροπές από τους ε, επιτρόπους Μογκερίνη, Μάλμστορμ και Μίμητσα. Βρισκόμαστε λοιπόν, όπως σας είπα, σε ύψος χρηματοδότηση περίπου 20 εκατομμυρίων για τα συνοδευτικά μέτρα. Ε, θα ακολουθήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη η σωστή ενημέρωση και θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και βεβαίως οι αντιπροσωπείες οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από αυτά τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων όλοι θα παραμείνουν ενημερωμένοι και θα δράσουν κατά τα επόμενα έτη. Είμαστε έτοιμοι βέβαια για να συνεχίσουμε και να συζητάμε και να παρακολουθούμε την πρόοδο στις διάφορες επιτροπές. Ευχαριστώ. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει τώρα το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, αναφερθήκατε στα πέντε κεφάλαια των συνοδευτικών μέτρων. Ε, καλό είναι βεβαίως κάποιος να έχει ε, κάποιος ο οποίος έχει γράψει ε, μια νομοθεσία στη συνέχεια να λογοδοτεί 3,5 χρόνια μετά για την εφαρμογή της. Εδώ έχουμε επικεντρωθεί σε ένα σημείο πρέπει οι εταιρείε να προωθήσουν ε, υπεύθυνη εξόριξη είναι βασική δέσμευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο όσα πρέπει να έχουν πραγματικά υπεύθυνες πρακτικές από τις επιχειρήσεις, ε, από τους επεξεργαστές, να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στην ετήσια συνάντηση του φόρουμ του ΩΣΑ, όπου προείδρευσα εγώ το πρόγραμμα των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων και που προτιμάζεται και η ατζέντα για το φόρουμ. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να συζητήσουν μεταξύ του ε, διάφοροι εμπλεκόμενοι φορεί. Θα θέλαμε λοιπόν τα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν ε, στι συναντήσει μα 19 με 24 Απριλίου, ε, σαν ένα μίνι νταβό κατά κάποιο τρόπο για υπεύθυνη αλυσίδα εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τι εξορίξει θα μάθετε έτσι απευθείας από την πηγή κάποια πράγματα από τις κυβερνήσεις, από την κοινωνία των πολιτών και από τις ίδιες τι επιχειρήσεις. Το φόρουμ μας έχει βοηθήσει να διαμορφώσουμε και μια σειρά από συγκεκριμένε πρωτοβουλίες επιτόπου ε, λύσεις ε, για τις περιοχές συγκρούσεων καθώς για την εξόριξη κασίτερου ε, και στο φόρουμ αλλά και στο διάλογο με την σε ό,τι αφορά τις, με, τις χώρες παραγωγής, επεξεργασίας και κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω εδώ πέρα ε, την ε, πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε από την κυρία Ράτσο. Ε, έχουμε αναλάβει το θέμα της υπεύθυνη ε, εξόριξη από τι περιοχέ συγκρούσεων. Στην Κίνα υπάρχουν πλέον κάποια, κάποιες προδιαγραφές που βασίζονται στι κατέσεις γραμμέ του ΩΣΑ και βασίζονται και στην υποστήριξη τη δική μα προ την ΩΣΑ έτσι ώστε να έχουμε ε, μία μετάφραση αυτών των στοιχείων ε, στην Κίνα και η Ινδία σιγά σιγά δεσμεύεται σε επίπεδο ΩΣΑ σε ό,τι αφορά την εξόριξη που οδηγεί στα σε κάποια κοσμήματα, στην παραγωγή κοσμημάτων, αλλά και στην εξόριξη πολύτιμων λίθων. Ε, υπάρχει μια υποστήριξη σε εθνικό, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο ε, εκ μέρους του ΩΣΑ. Ε, υπάρχει η περιφερειακή διάσκεψη για την εξόριξη και την πιστοποίηση. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την εξόριξη μικρής κλίμακας ε, την κοινωνία των πολιτών στην ακτή Ελεφαντοστού, στην Πουρκίνα Φάσο. Η κυρία Μακάβα αναφέρθηκε προηγουμένω και στο σχέδιο το οποίο προετοιμάζουμε με την ε, Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Για να είμαι όμως απολύτως ειλικρινής μαζί σας ε, στην ε, μηχανισμοί πιστοποίησης διεθνώς θα απαιτήσουν συνεχή δράση και από τις κυβερνήσεις. Θα πρέπει αυτά τα πιστοποιητικά να γίνουν όλο και πιο αποδεκτά ε, ήδη στην βάση της ε, αλυσίδας. Έχουμε ήδη στοιχεία τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν την προσπάθεια που κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Να αναφερθώ σε ένα στοιχείο στο τέλος του έτους ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, ζήτησε ε, να ενημερώνει η κυβέρνηση της, κεντρικής, της Δημοκρατίας Κεντρικής Αφρικής ό,τι αφορά τις εξαγωγές και στην τελική έκθεση από την ομάδα πυρογνωμόνων των ΗΠΑ γίνεται αναφορά σε κάποιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά την, ε, το λαθρεμπόριο που προκύπτει μετά από κατόπιν πρωτοβουλίας αυτής ε, είμαστε πριν από, πριν ένα χρόνο το 2017 ε, όπου τρία μέλη της Επιτροπής μας ε, μεταξύ των οποίων μία Σουηδή συνάδελφος ε, έχασαν τη ζωή τους σε μια επίσκεψη στην Κατάγκα προς τον Μπουρουντή. Ε, από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί να κάνουμε τη διαφορά χάρη στη due diligence αυτό αποτελεί μέρος και της, του κανονισμού του Συμβουλίου 90% του επεξεργασμένου χρυσού, ε, του ε, ε, μετάλλων που έχουν επικοινωνήσει αντικείμενο τήξης, όπως το ταντάλιο, να καλύπτονται. Τέσσερις, ε, τέσσερις, τέσσερα χρόνια για αυτά τα τρία τι, για αυτά τα, αυτά τα τρία μέταλλα ε, έχουν οδηγήσει ε, σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για χιλιάδες, πάνω από 100.000 οικογένειες. Βεβαίως η πραγματική ε, πρόκληση, μία από τις προκλήσεις, είναι ε, το λαθρεμπόριο χρυσού, διότι το 100% περίπου αυτού του λαθρεμπορίου φεύγει από την Κεντρική Αφρική χωρίς καμία ανείχνευση. όχι από την Κεντρική Δημοκρατία της, της ε, ε, Αφρικής, αλλά από το Κονγκό. Έγινε αναφορθά προηγουμένως στο GSP+. Αυτό αποτελεί μέρος ε, ε της εργαλειοθήκης για την καλή κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει για το due diligence. Πρέπει να υπάρχουν συνοδευτικά μέτρα. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά τα ευρύτερα ζητήματα διακυβέρνησης βασίζονται στην υποστήριξή βασίζονται στην δυνατότητα επιρροή που έχει η ΔΕΦΚΟ στι εν λόγω χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Θα ήθελα πραγματικά να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας και συγκεκριμένοι και να θέλετε ερωτήματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους επίσης. Έχουμε 15 λεπτά για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσαμε να λάβουμε πληροφορίες ε, ε σε αυτήν την επιτροπή ε, και να τα αφήσουμε για την Ολομέλεια. Εν περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την, την επερχόμενη μεταρρύθμιση της σχετικής οδηγίας για τη χρηματοδότηση και τη νέα ε, νομοθεσία την ενδεχόμενη για, υπερ, για υποχρεωτική due diligence. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη μπορεί να μας δώσει κάποιες ενδείξεις για τη διαδικασία αναθεώρησης της ε, οδηγίας ε, σχετικά με τις αναφορές για τα μη οικονομικά ζητήματα. Αυτό είναι σημαντικό για το θέμα του due diligence και βεβαίως συνδέεται και με την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι στην κυρία Ράτσο ήταν η η πρώτη ερώτηση, η Γιούντιτ Σαρχεντίνη. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να απευθυνθώ στον κατάλληλο. Βοηθήστε με κι εσείς κύριε Πρόεδρε για να μου πείτε ποιος είναι ο κατάλληλος απαντήσει. Διάβασα το με τη δράση για τις πρώτες δραστηριότητε των συνοδευτικών μέτρων και χαίρομαι που έχουμε πια τέτοιο φυλάδιο, τέτοιο δελτίο γιατί ε, όταν διαβάσαμε το 2014 την ανακοίνωση και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι μπορεί να είναι τα συνοδευτικά μέτρα, ουσιαστικά σκεφτήκαμε ότι το καλύτερο είναι να στηρίξουμε τις ε, χώρες της περιοχής των μεγάλων ε, λιμνών να αναπτύξουν περισσότερο την μεταξύ τους συνεργασία. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια και φαντάζομαι ότι κάποιος, ίσως από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, θα είναι ο αρμόδιος για να μου απαντήσει πώς τα σημερινά σχέδια και με ποιο τρόπο διαφέρουν από τα προηγούμενα. Είχαμε ένα σχέδιο πιλότο που χρηματοδοτήθηκε από την Ολλανδική κυβέρνηση, ε, η πρωτοβουλία πιστοποίησης για το εμπόριο κασίτερου, από κοινού και στη συνεργασία με συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για, τον υπεύθυνο αφοδιασμό ρηκτών από περιοχές συγκρούσεων, που επίση ε, το στηρίζει η Ολλανδική κυβέρνηση και σίγουρα πολλές εταιρείες αναμειγνύονται ε, σε αυτό το σχέδιο. Οπότε έχουμε αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Αλλά θα ξεπεράσουμε αυτή τη στάση, την πιλωτική φάση δηλαδή για την πιστοποίηση ορυκτών και μεταλλευμάτων ε, για εξαγωγή. Αυτό θέλω να καταλάβω. Οπότε θα περάσουμε στην επόμενη φάση μετά το πιλωτικό σχέδιο. Φαντάζομαι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η πρόταση, γιατί μιλάμε για 9,3 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 5,3 προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άκουσα 20 εκατομμύρια να αναφέρετε εσείς. Μπορείτε να μου παρουσιάσετε το σύνολο του πακέτου, γιατί τα συνοδευτικά μέτρα δεν φαντάζομαι να αφορούν μόνο το πιλωτικό σχέδιο για την πιστοποίηση που ήδη έχει ε, μάλλον εφαρμοστεί. Επίσης, τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε κι εσείς ε, για τον διαγωνισμό για τα δημόσια αγαθά ε, και τη σχετική νομοθετική διάταξη πώς θα εφαρμοστεί αυτή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης έχουμε και τις κατευθυντήριες ε, αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα αυτά. Και εκεί περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα άσκηση ενδικών μέσων, η επιβολή του νόμου, ε, διεκδίκηση κάποιας ε, διόρθωση αποκατάστασης. Πώς θα ληφθούν υπόψη στις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές και οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους τρεις καλεσμένους μας, τους εκπροσώπους ε, των δύο Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, θα πρέπει να δούμε όχι μόνο τα τεχνικά αλλά και τα πολιτικά ε, θέματα που είναι επίσης πολύ σημαντικά γιατί αφορούν και την ε, πολιτική και οικονομικο-κοινωνική κατάσταση αυτών των χωρών που βρίσκονται σε συγκρούσεις. Και επίσης θα πρέπει να περάσουμε ίσως σε μια πιο απτή, συγκεκριμένη και ίσως και ταχύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Εξού και η, πρώτη μου ερώτηση προς την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έχετε επίγνωση της επιτακτικής ανάγκης της επιτάχυσης αυτής της διαδικασίας, ακόμη και αν επίσημα ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόνο την 1η Πρώτου 2021. Δεν πρέπει παρόλα αυτά να επισπευστεί η διαδικασία. Δεύτερη ερώτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Έχουμε το εχειρίδιο και την βάση δεδομένων του κανονισμού. Πολύ σημαντικά στοιχεία για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δομές για την εφαρμογή του κανονισμού. Οπότε, α, τι γίνεται με τα αντίστοιχα εγχειρίδια και τις βάσεις δεδομένων, σε τι φάση βρίσκονται προκειμένου να, εφαρμοστεί, να βοηθήσουν την έμπρεκτη εφαρμογή του κανονισμού για τη δέωση επιμέλεια. Επίσης, από τη Γενική Διεύθυνση, στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τα συνοδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν και κάποια ενάυσματα, είπατε, κάποια κίνητρα. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα αρκεί να λέμε ότι απλώς ε, παροτρύνουμε τους ε, διαφερόμενους φορείς για τη διαδικασία ή δίνουμε κάποια κίνητρα. Εδώ υπάρχουν και κάποιες δεσμευτικές διατάξεις, κάποια υποχρεωτικότητα. Τι συγκεκριμένα συμμετευτικά μέτρα ε, επεξεργάζετε εσείς και τέλος για τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΠΑ Εθνών. Έχουμε και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για τη Διεθνώς Δεσμευτική Συμφωνία για την εταιρική ευθύνη ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι συναφές ε, και με το συγκεκριμένο κανονισμό. Πώς ε, συμβάλλεται ή στηρίζεται τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις που γίνονται στη Γενέβη. Θα μιλήσω γερμανικά για να ξεκουραστεί λίγο και η Γερμανή διερμηνή. Και έχω μία πολύ σύντομη ερώτηση. Επειδή ήμασταν πρόσφατα στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και διαπιστώσαμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διαμαντιών και του χρυσού ε, είναι αντικείμενο λαθρεμπορίου και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η σύγκρουση διότι οι ένοπλοι έχουν υπό την κατοχή τους όλα τα χρυσορυχεία κυβέρνηση τίποτα. Εμένα λοιπόν με ενδιαφέρει το εξή. Ε, εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση πώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κεντροαφρικανική δημοκρατία. Γιατί αν δεν υπάρχει έλεγχος στα ορυχεία και κυρίως στα χρυσορυχεία είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστούν οι συγκρούσεις. Ε, Τρεις ε, πολύ σύντομες ερωτήσεις θέλω να κάνω και οι τρεις απευθύνονται στην Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση. Η Κομισιόν ενθαρρύνει εταιρείε που καλύπτονται από τον κανονισμό να αρχίσουν να εφαρμόζουν την διαδικασία δέουσας επιμέλειας και πώς το παρακολουθεί. Δεύτερον, όσον αφορά ε, την εθελοντική δέουσα επιμέλεια, η Κομισιόν ε, ελέγχει το πώς αντιμετωπίζεται αυτές τις εταιρείε και πώς μπορούν να συγκριθούν όλα αυτά με τις οδηγίες του ΣΑ κατόπιν σχετικά με την σωστή εκμετάλλευση. Πώς προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε χώρες υψηλού κινδύνου ενώ παράλληλα να βελτιώνεται και η οικονομική και πολιτική κατάσταση των ε, γηγενών. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα σε αυτό τον γύρο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει δύο λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ τους συμπρόεδρους. Την τελευταία ερώτηση δεν κατάλαβα. Ίσως χρειαστεί να την επαναλάβετε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σχέδιο για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, είμαστε ακόμη σε προπαρασκευαστική φάση αυτού του πιλωτικού σχεδίου. Τώρα αναπτύσσουμε αυτό το σχέδιο από κοινού ε, με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε για την Κεντροαφρικανική δημοκρατία ε, για το χρυσό και τα διαμάντια. Δεν ξέρω ποιο, ποιο είναι το ποσοστό λαθρεμπορίου διαμαντιών από την Κεντροαφρικανική δημοκρατία. Πάντως έχουμε ένα σημαντικό σχέδιο που επεξεργαζόμαστε για το θέμα αυτό εν ώψη και της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018 στη διαδικασία του Κίμπερλι. Σε ό,τι αφορά την επιτάχυση της όλης διαδικασίας, Φυσικά, οι κατευθυντήρες γραμμές του ΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια δεν εμποδίζει τις ε, εταιρείε να εφαρμόσουν οικειοθελώ τη δέουσα επιμέλεια, γιατί όλοι γνωρίζουν πόσο σοβαρά είναι αυτά τα θέματα και στο Κονγκό. Και σε ό,τι αφορά ε, τις ερωτήσεις κυρίας Αρχεντίνη για την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τα υπεύθυνα ορυκτά, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ. Σε ό,τι αφορά τους κλειστούς αγωγούς, όλοι γνωρίζουμε τα όρια τους ε, και η Ολλανδική κυβέρνηση γνωρίζει τα όρια τέτοιου είδους σχεδίων του κλεισίματος τέτοιων διάβλων και φαντάζομαι ε, δεν θα επαναληφθεί αυτό το θέμα από την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τα υπεύθυνα ορυκτά. Σε ό,τι αφορά τι τις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Δύο τρίτα των κρατών μελών μέχρι στιγμής έχουν σχέδια δράσης για το θέμα αυτό. Και μάλιστα για να είμαστε ακριβείς στην απάντηση, δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερος με το θέμα αυτό. Πάντως, οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια του ΩΣΑ περιλαμβάνουν και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε, δεν υπάρχει καμία αντίφαση, καμία σύγκρουση μεταξύ των διαφορών κατευθυντηριών γραμμών και των κατευθυντηρίων αρχών του Ηνωμένου Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά τα νομικώς ε, δεσμευτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος και μάλλον αρμόδια είναι η Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο πρόσωπος τη ε, Γενική Διεύθυνση ε, αναπτυξιακή συνεργασία. Σίγουρα θέλουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση τη αλυσίδας εφοδιασμού από τη σήμερα. Δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση τη αλυσίδας εφοδιασμού μέσω διαγωνισμών ε, που θα δημοσιευθούν φέτο Η... Κάλεσμα για την υποβολή προσφορών. Τώρα να δούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Καταρχήν να διευρυνθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον αυτή τη βιοτεχνική βιοτεχνικής μικρή κλίμακο, να βοηθήσουμε την επισημοποίηση και επιστοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών με μεγαλύτερη σαφήνεια δικαίου μέσω οργάνωσης και επισημοποίηση των εκπροσώπων τη αλυσίδα εφοδιασμού και των διαφόρων φορέων ή παραγόντων σε όλη αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού. Οπότε Θέλουμε ε, να συνεργαστούμε με τους ενδιαφερομένους και να δούμε πώς θα, θα εφαρμόσουμε και την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για τα υπεύθυνα ορυκτά και πώς θα συνεργαστούμε με τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές που στηρίζουν τη διαδικασία, ώστε και με το... στα πλαίσια της ε, πολιτικής που έχουμε να υιοθετήσουμε ένα πιο ρωμαλαίο πλαίσιο, γιατί σίγουρα ε, τα σχέδια αυτά επηρεάζουν και τις τοπικές ε, κοινότητες, γιατί ήδη ε, είναι ορατές οι επιπτώσεις. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα γίνει εν μια νυχτή, πρόκειται για μια χρονοβόρα και μακρόπνοη διαδικασία. Όπως όμως είπε και ο εκπρόσωπος του ΙΕΔ, δεν μιλούμε μόνο για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ, αλλά και για τις προδιαγραφές της Διεθνούς Οργανούς Εργασίας και άλλες προδιαγραφές που θα καταστήσει τον κλάδο αυτό όσο πιο βιώσιμο γίνεται. Πάντως θέλουμε συνεργασία μαζί σας ώστε την επόμενη διετία να δούμε ποιες είναι οι επιτόπου δράσεις μας και η έμπρακτη εφαρμογή αυτών των πρωτοβουλειών στις πιο ευάλωτες περιοχές και χώρες. Η κυρία Ράτσο. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσω κάποιες πιο διεξοδικές πληροφορίες γιατί μας ρωτήσατε για την προετοιμασία Έχουμε προχωρήσει αρκετά στα θέματα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τις ε, χώρες μέλη και τις ε, ελέγχους εκ των ε, υστέρων και μάλιστα το εγχειρίδιο κανόνων που μας είπατε, μας ρωτήσατε, αυτό το εγχειρίδιο το συζητούμε ήδη με τα κράτη-μέλη και μάλιστα θα έχουμε μια συνάντηση των εμπειρογνωμόνων. Μάλιστα προσκαλέσαμε εκεί και το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Θα γίνει στις 9 Μαρτίου ε, η συνάντηση των εμπειρογνωμών και καλέσαμε και εκπροσώπους των αρμοδίων, χωρών, των αρμοδίων αρχών των χωρών μελών. Έτσι κύριε Βίνκλερ, θα βοηθήσουμε τις αρμόδιες αρχές ε, σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί και οι αρμόδιες αρχές είναι έτοιμα τη ε, διαδικασίας, μπορούν να την επηρεάσουν και μπορούν με την ανταλλαγή απόψεων και με τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή να αλληλοβοηθηθούν και να εκμεταλλευτούν ο ένας τα επιτεγμάτα του άλλου. Σε ό,τι αφορά το non-financial reporting, κυρία Χάουταλα, ήδη από πέρυσι είχαμε μια εφαρμογή που καλύπτει τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων ή συγκεκριμένα την ε, ειδική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από τις μεγάλες εταιρείες υπό το πρίσμα και της δεούσας επιμέλειας. Υπάρχει δηλαδή αυτή η υποχρέωση ήδη. Τώρα τι κάνουμε για να εθαρρύνουμε τις ε, εταιρείε και ανάντι και κατάντι να εφαρμόσουν ε, νωρίτερα την ε, υποχρέωση της δέωσης επιμέλειας και πριν την 1η του 2021 που θα αρχίσει να εφαρμόζεται επίσημο ο κανονισμός τους. Εθαρρύνουμε λοιπόν να εφαρμόσουν πιο νωρίς αυτή τη δεωση επιμέλεια και μάλιστα για τις εταιρείε κατάντι συγκεκριμένο μέτρο θα είναι η πλατφόρμα της διαφάνειας που πρόκειται να ξεκινήσει φέτος ε, ώστε να μπορέσουν και οι εταιρείε που βρίσκονται σε κατάντη να παράσχουν πληροφορίες για πρακτικές δέουσες επιμέλειες. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Είδατε και τις παρεμβάσεις των μελών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο ήδη από την προηγούμενη θητεία του. Είχαμε ζητήσει αυτό το μέτρο. Βεβαίως είναι χρειάζεται χρόνο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τέτοιου είδου μέτρα. Υπάρχουν ζητήματα διακυβέρνηση σε πολλέ από αυτέ τι χώρε ε, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ε, καθώ και ζητήματα διακυβέρνηση ε, στο δικό μα επίπεδο, από τη δική μα πλευρά. Ελπίζω να συνεχίσετε πάντω να ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωση, όταν προκύπτουν δυσκολίε, να μα το λέτε. διότι συχνά λέμε ότι κάτι είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει, δεν θα λειτουργήσει, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά με λίγη πίεση. Βλέπουμε τώρα ότι στην Κίνα και σε άλλες χώρες ε, υπάρχει μια βελτίωση και έχουμε εμείς ουσιαστικά ε, δείξει το δρόμο, έχουμε δημιουργήσει ένα μοντέλο το οποίο ακολουθείται πλέον παγκόσμια. Ελπίζω να συνεχίσετε να μα ενημερώνετε λοιπόν. Θα έχουμε μια συζήτηση με την, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιο θα είναι ο επίτροπο βέβαια στην Ολομέλεια. Ε, Σα ευχαριστώ πάντω πολύ. Να πω τώρα κάτι στου αδέλφους τη επιτροπή ΔΕΒΕ. Τέσσερι η ώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίασή μα. Θα πρέπει να περπατήσουμε όμω. PHS 4V001 είναι το, ε, στο κτίριο της, ε, της Λομέλειας, ε, ο κύπρος και το κύκλιο δηλαδή, στον πέμπτο όροφο. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστώ Λίντα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που ήσασταν μαζί μας. Είναι μια καλή πρακτική αυτή, είναι να ακολουθούμε μια κοινή προσέγγιση δηλαδή και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ε, τις επιθυμίες μας. Θα έχουμε άλλη μια επικοδομητική συζήτηση τον επόμενο μήνα και φαντάζομαι ότι αύριο η κάθε επιτροπή θα εγκρίνει τις προφορικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.